So, liebe καλησπέρα σας. Ε, ε, καλημέρα σας στη συνεδρία σήμερα το πρωί τη Επιτροπής μας μετά από τον μαραθώνιο των ψηφοφοριών εχθές. Έχουμε ακόμη δύο βασικά θέματα στην ημερήσια διά, ημερήσια διάταξη τις ε, εκπομπές ε, τις βιομηχανικές ε, και τις εκπομπές για τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών θα σας μεταδοθούν γραπτών, οπότε θα ασχοληθούμε τώρα με τις βιομηχανικές εκπομπές, ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρήπανσης ε, με εισηγήτρια τη Χόλγκερ, τον Χόλγερ Κράμερ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Νομίζω ότι σχετικά με την οδηγία των βιομηχανικών οδηγών έχουμε ε, ένα μεγάλο εργοτάξιο που μας περιμένει όπως ε, και εχθές με τα τρόφιμα και ελπίζω ότι θα έχουμε πολλή δουλειά ως το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε την πρώτη ανάγνωση ε, αφού το προηγούμενο κοινοβούλιο είχε ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση κατά τρόπον ώστε να έχει επαρκή χρόνο και το Συμβούλιο να διατυπώσει τις θέσεις του και να μπορέσουμε ε, να καταρτήσουμε νέους κανόνες επιτροπολογίας ε, κατόπιν ε, της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας και έτσι τώρα ξεκινούμε τη δεύτερη ανάγνωση. Θα ήθελα να σας και εντάχει γιατί ίσως δεν έχουν όλοι ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα για να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται ε, για ε, περίπου 50.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες αφορούνται στην Ευρώπη σχετικά με ε, τις επιταγές οι οποίες θα εφαρμοστούν για αυτές τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Και ξέρετε ότι ήδη υπάρχει μια οδηγία η οποία όμως δεν εφαρμόζεται σωστά. Και γιατί αυτό διότι ο ουσιαστικός στόχος της οδηγίας είναι η ε, χρήση συγκεκριμένων τεχνικών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και ε, δυστυχώς με την ισχύουσα οδηγία διαπιστώνουμε ότι η ευελιξία την οποία χρειαζόμαστε ε, επιγόντως στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη δεν ε, καλύπτονται σωστά από την ισχύουσα νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχει μία ευελιξία την οποία χρησιμοποιούν προς όφελός τους οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δεν εφαρμόζουν σωστά την ε, ε, τωρινή οδηγία όσον αφορά την χρήση των βελτίστων ε, πρακτικών. Στην πρώτη ανάγνωση είχαμε προσπαθήσει να βρούμε ένα τρόπο με τον οποίο θα ε, εξετάζαμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη χρήση της υπαρχούσης νομοθεσίας και είχαμε αναφερθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασφαλείας το οποίο είχε καταρτιστεί στις Βρυξέλλες και ε, το οποίο τελικά δεν μπορούσε κανείς ε, να αντιπαρέλθει και στην πρώτη εφόσον θα εφαρμοζόταν και ε, ευχαριστώ για την πρώτη ανάγνωση και για τους συναδέλφους που με βοήθησαν τότε αλλά εξετάζοντας το αποτέλεσμα είδαμε ότι το Συμβούλιο δεν κατάλαβε την ιδέα μας ουσιαστικά την απέρριψε και η θέση εάν την εξετάσουμε τώρα δεν ισχύει όπως εις ε, την περιβαλλοντολογική νομοθεσία αλλά θεωρείται σαν μία εξαίρεση. Δηλαδή υπάρχει μία θέση του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση και μία θέση του Συμβουλίου οι οποίες είναι διαμετρικά αντικρουόμενες και πρέπει να οδηγηθούμε σε μία νομοθεσία η οποία θα μπορέσει να βελτιώσει την ισχύουσα κατάσταση σχετικά με αυτή την οδηγία. Εν ώψη λοιπόν αυτής της ε, καταστάσεως, ε, χωρίς να θελήσω να ε, περί προσπάθησα να λάβω υπόψη ε, το τι ε, είχε συμβεί, δηλαδή ε, να θεωρήσω ότι οι αρχές δεν έπρεπε να θεωρηθούν δεδομένες, έπρεπε να τροποποιηθούν για να υπάρχει τουλάχιστον ένα κατώτατο όριο εφαρμογής. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να στηρίξετε την άποψη αυτή. Θα μου πείτε γιατί χρειαζόμαστε κατώτατες προδιαγραφές εφόσον υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και ορισμένοι θα πούν αυτές είναι γερμανικές ιδέες οι οποίες προσπαθούν να εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη αλλά νομίζω θα είναι προς όφελος όλων εάν κάτι τέτοιο καταρτιστεί το οποίο να επιτρέψει να υπάρχει μία ανταγωνιστικότητα μεταξύ ίσων πράγμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή χώρες οι οποίες προχωρούν καλά και χώρες που δεν κάνουν τίποτα. Άρα οι κατώτατες προδιαγραφές θα είναι ένας τρόπος καλύτερης εφαρμογής των διαθεσίμων τεχνικών. Και ε, ουσιαστικά ε, λέγεται το εξής η πρόταση μου για την έκθεση αυτή τώρα ε, προβλέπει ε, τα συμπεράσματα από τις διαθέσιμες τεχνικές να εφαρμοστούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει μία έκθεση η οποία ιδίως θα ερευνήσει δύο κριτήρια. Δηλαδή, καταρχήν, πώς προχωρά η εφαρμογή των διαθεσίμων τεχνικών τώρα και πώς επηρεάζεται το περιβάλλον και μετά από αυτό να αποφασίσουμε εάν χρειάζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ε, αν ε, ε, απέχουν πάρα πολύ από τα ισχύοντα. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε μία κατάσταση η οποία να αναφέρεται στον συγκεκριμένο τομέα και να διατυπώνει ελάχιστες προδιαγραφές και το λέω πολύ σαφώς προσπαθώ να προσεγγίσω το Συμβούλιο διότι είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ένα άλλο βασικό θέμα το οποίο εμφανίζεται εδώ και ουσιαστικά θα σκιαγραφίσω τρία ουσιαστικά σημεία της εκθέσεώς μου και όχι όλες τις λεπτομέρειες διότι διαφορετικά θα μακρηγορήσω πάρα πολύ και θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στους αδέλφους να μας πούν τι σκοπεύουν να κάνουν. Ε, μιλάμε πάρα πολύ για τις εξαιρέσεις. Στο άρθρο 15 παράγραφος 4 μιλάμε που μπορούμε να αποκλείσουμε από τις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές. Και εδώ είμαι πεπισμένος ότι μπορεί κανείς να παρεκκλήσει ε, αν ε, ε, ε, αν χρησιμοποιήσει ορισμένες μεθοδολογίες διότι πιστεύω ότι οι βέλτιστες τεχνικές δεν είναι ουτοπία, δεν είναι επιστημονική φαντασία, δεν είναι τόσο δαπανηρές, αλλά είναι η ισχύουσα κατάσταση, δηλαδή το status quo της τεχνικής και δεν μπορεί κανείς να παρεκκλίνει ιδίως εάν ε, χτίζει νέες εγκαταστάσεις. Άρα αυτό το οποίο ήθελα ήταν από την πληθώρα των ε, εξαιρέσεων που υπάρχουν να μπορέσουμε να διατυπώσουμε ε, με μονομένες ε, αποκλειστικές εξαιρέσεις οι οποίες να βασίζονται σε αιτιολογημένες αποφάσεις. Όσον αφορά το τρίτο βασικό θέμα αυτής της οδηγίας πρόκειται για τις εγκαταστάσεις καταστάσεις ε, ε, των, ε, των εγκαταστάσεων καύσεως και εδώ υπάρχει η προσπάθεια να μειωθούν οι βλαβερές εκπομπές υπομορφή αερίων και εδώ το, στο κεφάλαιο 3 Τρία, προβλέπεται ένας τεράστιος κατάλογος εξαιρέσεων, προϋποθέσεις και συνθήκες υπό τις οποίες οι οριακές τιμές δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό δεν μας βοηθάει. Εάν προχωρήσουμε έτσι ε, μπορούμε να αφήσουμε την περιβαλλοντολογική νομοθεσία ως έχει διότι τότε το κάθε κράτος μέλος θα συνεχίσει να κάνει ό,τι, ό,τι επιθυμεί και θα ήθελα με την στήριξη όλων των ε, κρατών μελών να ε, επιτύχουμε ε, πολύ φιλόδοξους στόχους στην ποιότητα αέρα στην Ευρώπη μέχρι το 2020 και να έχουμε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών ιδίως όσον αφορά το μονοξίδιο του αζότου, το διοξίδιο του αζότου, το διοξίδιο του θείου διότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτές τις τιμές εάν ε, δεν ε, συζητήσουμε τις εξαιρέσεις αυτές. Μιλάμε και για τις ε, μετακινήσεις, τις μεταφορές, όπου έχουμε λιγότερες δυνατότητες επεμβάσεως με χαμηλό κόστος, αλλά μπορούμε με χαμηλό κόστος να βελτιώσουμε την κατάσταση της βιομηχανίας. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτύχουμε μια σημαντική πρόοδο τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Στην έκθεση έχω προτείνει πολύ ριζικά μέτρα και έχω ήδη ακούσει ορισμένα σχόλια από εκπροσώπους του Συμβουλίου και ορισμένων ενδιαφερομένων, δηλαδή έχω διαγράψει τα εθνικά μεταβατικά προϊόντα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ενιαία ικανοποιητική λύση. Δηλαδή τα Transitional National Plan, τα μεταβατικά εθνικά προγράμματα προβλέπουν ότι ε, ως όσοι έχουν μία άδεια πριν από το 2002 δεν χρειάζεται να επιτύχουν τους επιθυμητούς στόχους πριν από το 2020 και επίσης έχει διαγραφεί η ε, πρόβλεψη ότι οι μεγάλες εγκαταστάσεις εσωτερικής κάψεως δεν χρειάζεται να λάβουν ορισμένα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και οι παλιές εγκαταστάσεις ε, εσωτερικής καύσεως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους και ε, το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι μικρές ε, βιομηχανίες είναι ότι η μεγαλύτερη αντίσταση για τις πιο αυστηρές απαιτήσεις προέρχεται ακριβώς από τα κράτη τα οποία δεν μπορούν να πούν ότι έχουν μία ανταγωνιστική βιομηχανία. Δηλαδή αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι πρόκειται για χώρες που ε, είναι πολύ οπισθοδρομικές σχετικά με το επίπεδο της βιομηχανίας τους και αυτές είναι ακριβώς ε, που ανθίστανται ε, για την εφαρμογή των νέων τεχνικών ιδίως στις εγκαταστάσεις ε, μεγάλων κλιβάνων και ε, θα έπρεπε να ε, συγκεράσουμε τους στόχους όλων των ενδιαφερομένων, να εφαρμόσουμε τη διαθέσιμη τακτική και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στον τομέα αυτό τους, τη διαθέσιμη τεχνολογία διότι ξέρουμε ότι οι μανούβρες όπως λέγουν, μάλλον οι δυνατές κινήσεις είναι περιορισμένες και το λέω σαφώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι προβληματικό εάν η ε, τωρινή προεδρία προεξοφλεί την, κατάστα... το... την έκβαση πριν καν να διαπραγματευτούμε και, να... και λέει ότι πρέπει να πάμε σε ε, ε, διαμεσολάβηση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει μεν ε, να διαπραγματευτούμε, εγώ είμαι διαθέσιμος, αλλά θα πρέπει να καταλάβει και η άλλη πλευρά ότι στη δεύτερη ανάγνωση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μόνο αν ε, υπάρχει μία ισχυρή ε, θέση του Κοινοβουλίου που θα αντιπαραταχθεί στη θέση του Συμβουλίου και ε, το έχω συζητήσει με τους κοιόδης εισηγητές και των διαφόρων πολιτικών ομάδων λέγοντας ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε αυτό που κάναμε και στην πρώτη ανάγνωση δηλαδή θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια ευρεία συνένεση η οποία πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά αλλά θα επιτύχει το στόχο ότι δηλαδή θα αλλάξει κάπως το τοπίο ε, όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις μεγάλες εγκαταστάσεις ε, καύσης και για τις εξαιρέσεις. Νομίζω ε, θα παραμείνω εδώ και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Θα έχω επιπλέον την δυνατότητα στη συνέχεια να απαντήσω στις ερωτήσεις οι οποίες ενδεχομένως θα μου τεθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμα. Μας κάνατε μια καλή εισαγωγή σε ένα σημαντικό το θέμα της περιβαλλοντική πολιτική και τη περιβαλλοντική Νομοθεσία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η οδηγία αυτή υιοθετεί και το 1996, η αρχική οδηγία εννοώ. 15 χρόνια έχουν περάσει από τότε και η αναθεώρηση βρίσκεται επιτάπητο γιατί η Κομισιόν ε, παρατήρησε ότι δεν εφαρμόζεται σωστά η οδηγία αυτή. Η εφαρμογή της από τα κράτη-μέλη δεν είναι ικανοποιητική. Η καθαρότητα του αέρα είναι ένα υψηλό αγαθό, όπως και η καθαρότητα του νερού. Ξέρουμε τις επιπτώσεις που έχει αυτό στα παιδιά ιδίω και σε άλλους με ασθένειες των αναπνευστικού συστήματος. Το έχουμε συζητήσει πλειστάκι εδώ, στην Επιτροπή μας. Και βέβαια δεν είναι καλό να συζητάμε θέματα τα οποία δεν τηρεί μετά κανένας. και θα πρέπει να αποφασίσουμε προς τα που θα κινηθούμε. Έχουμε ένα κείμενο πάνω στο οποίο συζητάμε. Θα δώσω το λόγο στους συντανιστές και μετά στους υπόλοιπους. Για το ΕΛ η είναι η πρώτη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή ο οποίος ε, επιτελεί μεγάλο και πολύ σημαντικό έργο. Στάθηκε σε πολλά επιμέρους ζητήματα, στα οποία θα ήθελα να σταθώ και εγώ. Ως προς τις ε, μεταφορές, εγώ έχω εντελώς διαφορετική άποψη, γιατί νομίζω ότι ότι η Επιτροπή Μεταφορών εργάζεται για μείωση 20% την επόμενη δεκαετία και βελτίωση ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος μέχρι τώρα. θεωρώ ότι αυτός ο κοινό κατάλογος είναι ένας κατάλογος εξαιρέσεων και τίποτα άλλο. Διότι το Συμβούλιο ζητά την αιτιολόγηση των ενδεχομένων εξαιρέσεων που θα ζητηθούν. Πριν όμως μπούμε στα διάφορα σημεία, θα ήθελα να μην επανέλθουμε στο, στα ζητήματα της πρώτης ανάγνωσης, διότι έχουν αλλάξει τα συμφραζόμενα. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά τις εκλογές ε, είχαμε μία αλλαγή, μεγάλες ε, αλλαγές ως προς τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, κατά 50% και η κοινή θέση εγκρίθηκε χωρίς αντιγνωμίες μόνο τέσσερα κράτη απέσχουν. Ξέρουμε ότι διανύουμε μια οικονομική κρίση η οποία όλο ένα και επεκτείνεται. Γι' αυτό αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θεωρώ ότι το κείμενο του Συμβουλίου είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις και μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Θεωρώ ότι αυτός πρέπει να είναι ένας από τους στόχους μας. Θα ήθελα να σταθώ στο European Safety Net. Ας μην ξεχνάμε ότι το Συμβούλιο απέριψε αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασφαλείας και η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί έμπρακτα. Και αυτό για συγκεκριμένους λόγους. Διότι μας είπε η Κομισιόν ότι δεν υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη εργασία. Και δεν ξέρουμε και πού να βάλουμε αυτό το προσωπικό για να προβεί στις αναλύσεις, στις σωστές αναλύσεις για το επίπεδο εκπομπών για κάθε τομέα. Το European Safety Net είναι πολύ αποδοτικό στη Γερμανία, αλλά χρειάστηκαν 10 χρόνια μέχρι ότου συσταθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η εργασία θα μπορούσε ε, να παρατείνει, να αναβάλει για ακόμα μακρύτερα τους στόχους μας. Όταν ο κύριος Κράμερ λέει ότι χρειάζονται αναλύσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εμβαθύνουμε το όλο σχέδιο έχει δίκιο. Αυτό σημαίνει περαιτέρω καθυστέρηση. Αν θέλουμε να φτάσουμε στους στόχους μας, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ο πιο σύντομος δρόμος και η νέα εκδοχή του European Safety Net που απασχόλησε τον κύριο Κράμερ ορίζει ελάχιστες τιμές μόνο για ορισμένους τομείς δραστηριότητας που θα αποτιμηθούν από την Κομισιόν ανάλογα με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Θεωρώ ότι αυτή δεν είναι αποδοτική πορεία ή πλέον αποδοτική. Ε, βλέπω ότι η δεύτερη έκδοση οδηγεί σε πολλά προβλήματα. Καταρχήν, διάκριση κατά ορισμένων τομέων. Υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για ορισμένους τομείς, για άλλους όχι. Επίσης υπάρχει και διάκριση κατά ορισμένων κρατών μελών. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να αφήσει το όλο έργο στην Επιτροπή να αναγνωρίσει αυτούς τους τομείς και τα κράτη. Και υπάρχουν και καταχρήσεις και από τις επιχειρήσεις, διότι οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να μην ακολουθήσουν την οδηγία και έτσι η Επιτροπή να φτάσει στα ανάλογα συμπεράσματα. Θα ήθελα επίσης να ξέρω να μας πει η Επιτροπή ποιοι ενδεχομένως είναι αυτοί οι τομείς που θα εξατομικεύσει η Επιτροπή και κατά πόσο άλλαξε άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις αρχικές της ανακοινώσεις κατά την πρώτη ανάγνωση για να ξέρω κατά πόσο τώρα υπάρχουν ανοίγματα από την Επιτροπή και κατά πόσο σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή βλέπει τέτοιες αλλαγές έτσι ώστε να ακολουθήσει αυτή την οδό. Νομίζω ότι είναι επίγον το θέμα της επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων. Και αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι πρόκειται για έναν μακρύ δρόμο. Γιατί πολλά κράτη-μέλη είχαν ε, δυσκολίες να εφαρμόσουν το EPPC όταν άρχισε αυτή η διαδικασία το 2007. Και πρέπει να σας ε, υπενθυμίσω ότι δεν σημαίνει ότι δεν φτάσαμε σε απτούς στόχους. Εδώ έχω στοιχεία που δείχνουν τους απότερους στόχους της Ευρώπης των 27 σε σχέση με, τη, ε, με τις εκπομπές. Βλέπουμε ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την πορεία. Και η ευρύτερη οικονομική κρίση μας οδηγεί στο να αναλάβουμε μεγάλες ευθύνες, διότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις χώρες μας και να πούμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν ε, μία νομοθεσία που δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί και θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί έχετε υπερβεί το χρόνο σας κατά πολύ. Τελειώστε την πρότασή σας. Αυτό μόνο. Δεν μου το είπατε, δεν μου είπατε πόσα λεπτά είχα στη διάθεσή μου. Εντάχει λοιπόν, θα πρέπει να επιβεβαιώσω το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία ο εισηγητής αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ευελιξίας ως προς την οδηγία που ισχύει και θα πρέπει να υπάρχει και μία αντιστάθμιση, δηλαδή οι εξαιρεσει να αιτιολογούνται πλήρως. Γι' αυτό προτείνω και μία τροπολογία, σύμφωνα με την οποία τα κράτη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εξαιρεσει και να τις αιτιολογούν. Και τα μεταβατικά σχέδια είναι ουσιώδη. Δεν έχετε άλλο χρόνο, σας παρακαλώ, πρέπει να σας διακόψω. Έχουμε 20 ε, παρεμβαίνοντες, συν την Κομισιόν, συν τον εισηγητή. Άρα οι συντονιστές να έχουν 20 λεπτά συνολικά και 2 λεπτά ο κάθε άλλος ομιλητής. Βέστλουντ και αρχίζει και να τρέχει και ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κράμερ για την ε, πάρα πολύ καλή του έκθεση. Είναι θετικό που αναφέρεστε στην θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση γιατί ήταν μια πολύ καλή θέση με φιλόδοξες αλλά όχι ιδιαίτερα ακριβές λύσεις. Δεν μπορούσα να έχω αναλυτική συζήτηση με την ομάδα μου για το θέμα, αλλά θα συστήσω τα εξή. Το είπαν ήδη κάποιοι από τους Η εφαρμογή της οδηγίας αυτής δεν ήταν επαρκής και αυτό είχε συνέπειες για την, το περιβάλλον και για την δημόσια υγεία. Και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για πολλές επιχειρήσεις ε, να ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει υψηλές προδιαγραφές ε, για την προστασία του περιβάλλοντος, ότι μπορούν δηλαδή να ε, εφεύρουν νέες πράσινες τεχνικές που θα μπορούν να τις εφαρμόσουν κιόλας. Αυτό οδηγεί σε κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα. Συγκεκριμένα, έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο, ακρι... πιο αυστηρά κριτήρια για τις εγκαταστάσεις καύσης και όσον αφορά τις εκπομπές. Ένα από τα κριτήρια που προτείνει ο κύριος Κράμερ ε, το, στο 15.4 γάμα μου φαίνεται ότι είναι κάτι που ήδη εφαρμόζεται μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης διαδικασίας της Σεβίλιας. Και γι' αυτό μου φαίνεται ότι είναι περιττό να το ξανααναφέρουμε. Θα επικαλύπτουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Οι παλιές ε, εγκαταστάσεις θα πρέπει να επιτρέπουν ε, κάποιες εξαιρέσεις. Τώρα βέβαια οι εξαιρέσεις για τις μεγάλες εγκαταστάσεις ε, καύσης δεν ξέρω γιατί αυτές ε, αφορούν το 90% των εκπομπών διοξιδίου του θείου και μια εξαίρεση θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές. Η Βρετανική κυβέρνηση που απολόγισε ε, ότι εάν εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις θα υπάρχει μια αύξηση του 2% για το διοξείδιο του άνθρακα και, του, του θείου και για τα οξύδια του αζότου και 4% για τα σωματίδια και γι' αυτό χαίρομαι που θέλουμε να διαγράψουμε την εξαίρεση για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Και επίσης όμως δεν συμφωνώ να έχουμε εξαίρεση για τις ε, εγκαταστάσεις 20 με 40 ΜΒ. Θεωρώ σημαντικό να μην ξεχνάμε ποτέ ότι υπάρχει πάντα ένα κόστος. Εάν δεν κάνουμε τίποτα θα πληρώσει το κόστος ο φορολογούμενος γιατί θα ανεβεί το κόστος της προστασίας υγείας ή της ε, θεραπείας ε, ασθενειών και μάλιστα εκείνοι που θα πληγούν ιδιαίτερα θα πληρώσουν με την ίδια τους τη ζωή. Αυτό το κόστος θα πρέπει επίσης να το έχουμε υπόψη μας. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν θα πληρώσει ο Ριπένον και γι' αυτό ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μια ισχυρή θέση του Κοινοβούλιο. Θα πρέπει, Πρόεδρε, να έχουμε κατ' ουσία όμως συζήτηση για το θέμα της, προστασίας ε, του περιορισμού του χρονογόρευσης. Γιατί στις περισμένες συζητήσεις πάντα όταν έφτασαν να πάρουν το λόγο οι σοσιαλδημοκράτες δεν είχαν τόσο λόγο όσο οι άλλοι. Πρόεδρος, ναι, θα βρούμε κάποια ισορροπία γιατί δεν είχα φανταστεί ότι η πρώτη παρέμβαση θα ήταν τόσο μακρά. Μπασέκοτ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χόλογκαρ Κράμερ για την εργασία του μέχρι στιγμή για το θέμα αυτό. Είναι τεράστιο θέμα και είναι καλό που ξεκινάμε πια τη δεύτερη ανάγνωση. Ε, έχει πιάσει το πλήρωμα του χρόνου. Θα παραμείνω στα τέσσερα λεπτά που μου είπατε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Ναι, αυτό που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι αν κοιτάξει κανένα στη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη, βλέπει ότι υπάρχουν τεράστιε διαφορέ για την εφαρμογή τη οδηγία αυτή. Ε, αν δει κανένα τι γίνεται στην Ολλανδία και στη Γερμανία σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπει ότι υπάρχουν τεράστιε διαφορέ μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων, χωρί να υπάρχει κανένα λόγο διότι η τεχνολογία είναι ίδια. Όταν συζητάμε λοιπόν για εσωτερική αγορά που είναι σημαντική για όλε τι πολιτικέ ομάδε. Θα έλεγα ότι ακριβώς λόγω της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα. Αυτή η οδηγία λοιπόν είναι σαφές ότι θα πρέπει να ξαναδιατυπωθεί για να οδηγήσει σε ίσες ευκαιρίες μεταξύ όλων των κρατών μελών. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό στη νέα αυτή διατύπωση οι δυνατότητες εξαίρεσης να ελεγχιστοποιηθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, να φροντίσουμε έτσι να λειτουργήσει η αγορά και να ξαλείψουμε τις άδικες διαφωνίες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι περίεργο ότι και οι εταιρείε ζητάνε για πιο αυστήρα, να υπάρχουν πιο αυστηρά μέτρα. Και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε. Κάτι άλλο. Συζητάμε το θέμα του κόστους Κάτι τη εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογιών. Αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι και οι ευκαιρίες που προσφέρονται για καινοτομία και τα κίνητρα για την έρευνα και την ανάπτυξη <clears throat> είναι πολύ σημαντικά και άμα δείτε και τις δυνατότητες απασχόλησης στην οικολογική βιομηχανία είναι επίσης σημαντική. Υπάρχουν δηλαδή και πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο με ανεκτήματα. Και άμα δείτε την αξιολόγηση των επιπτώσεων επιπτώσεων της Κομισιόν και δείτε τις εξοικονομήσεις για την υγεία, 65 δις ευρώ ανά έτος θα εξοικονομηθούν το 2020 λόγω της εφαρμογής οδηγίας αυτής. Και το κόστος, το όφελος μάλλον για τις επιχειρήσεις θα είναι 20 πλάσιο από το κόστος της συμμόρφωσης με την οδηγία. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. υποστηρίζουμε λοιπόν τον εισηγητή, το ξέρει βέβαια, που προσπαθεί να μειώσει τον ρυθμό των εξαιρέσεων και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι η διαγραφή των μεταβατικών εθνικών ε, προγραμμάτων για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Εδώ θα υποστηρίξουμε απόλυτα τον εισηγητή. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω ενδυνάμωση του κειμένου όταν αφορούν ε, τους ε, όρους για εξαιρέσεις θέλουμε να αφορά αυτό μόνο τις υψίουσες εγκαταστάσεις, να υπάρχει χρονικός περιορισμός και να επιτρέψουμε γενικά τις εξαιρήσεις ε, ούτως ώστε να μην υπάρχει ένα όφελος, ε, μάλλον μια εξαίρεση στην περίπτωση που υπάρχει όφελος της μη συμμόρφωσης και θα πρέπει αυτό να υπολογιστεί ένα του κόστους για το περιβάλλον. Καλή οδηγία, θέλουμε όμως να ενδυναμώσουμε το κείμενο γιατί μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και ωφελεί τη δημόσια υγεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους πολίτες. Τέσσερα λεπτά πρόεδρε. Very sharp. Yeah, yeah. So Martin Λοιπόν, ο Μάρτιν Κάλλαν. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του και για την συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητής διότι υπήρξε πάρα πολύ ε, χρήσιμη. Όσον αφορά την έκθεσή του και τα θέματα που θίγει υπάρχουν ορισμένα καλά στοιχεία και συμφωνώ μαζί του όσον αφορά την διαγραφή ε, του, ε, του σκεπτικού ε, για την εμπορία των εκπομπών. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ικανοποιητικό τρόπος για να μειωθούν οι εκπομπές. Συμφωνώ με την τροπολογία 14 για τα έγγραφα που θα δημοσιεύονται και δεν είναι σωστά σημεία αναφοράς και επίσης όσον αφορά την δημοσίευση σε όλες τις γλώσσες όσες που χρειάζονται. Αυτά όμως τα οποία δεν συμφωνώ και δεν θα εκπλαγεί είναι η τροπολογία 16 και 17. Δηλαδή ε, η επαναφορά του ε, Ευρωπαϊκού Δίκτυου δικτύου ε, ασφαλείας το οποίο προτείνει διότι εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσω συναποφάσεως και όχι μέσω επιτροπολογίας όπως προτείνει. Πέραν αυτού Έχω δυσκολίες όσον αφορά την, την τροπολογία που αλλάγει τα κριτήρια για τις εξαιρέσεις και περιορίζει στις εξαιρετικές συνθήκες, πράγμα με το οποίο δεν συμφωνώ. Με ανησυχεί ιδιαιτέρως η διαγραφή της των μεταβατικών εθνικών προγραμμάτων. Αντιλαμβάνομαι την αποψή του, δεν συμφωνώ μαζί του και πιστεύω ότι και σε πολλά κράτη-μέλη με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε ε, ε, εισαγωγή μέτρων ε, εκτάκτου ανάγκης για να καλυφθεί το κενό και η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, μεγάλων εγκαταστάσεων καύσεως οι οποίες δεν θα μείωναν τις εκπομπές. Τέλος, η τροπολογία 38 σχετικά με τη διαγραφή ε, της εξαιρέσεως του περιορισμένου χρόνου λειτουργίας δεν με βρίσκει σύμφωνο και θα ήθελα να ξανασκεφτεί την πρότασή του σε αυτό το θέμα. Τέλος θα πρότεινα ε, να υπάρξουν τροπολογίες σχετικά με ε, την ε, μεταβατική τεχνολογία επεμβάσεως και θα υποβάλω τροπολογίες από αυτού του θέματος για εξέταση από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, παρόλο που δεν συμφωνώ ε, με διάφορα θέματα και μάλιστα καθόλου όσον αφορά τις γενικές ιδέες της εκθέσεως δέχομαι το γενικό πνεύμα του εγγράφου και ε, το να επανέλθουμε στις θέσεις της πρώτης ανάγνωσης και συμφωνώ με τον εισηγητή για την ανάγκη να περιορίσουμε τις εκπομπές από τις βαριές βιομηχανίες και ιδίως αυτές που καίουν βαριά καύσιμα. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να προσφύγουμε σε ε, μέσα της αγοράς ε, ως προς τα, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θείου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, αφαιρέσουμε τη μνήμα σε αυτή τη δυνατότητα. Από όσο κατανοούμε, θα πρέπει να υπάρχει μία, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου γιατί είδαμε ότι μέχρι το 2005 το ευρωπαϊκό σχήμα ανταλλαγής εκπομπών δεν ήταν αποδοτικό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία ε, ρύθμιση όλων των εκπομπών παρά να διευρύνουμε το πλαίσιο σε άλλα είδη εκπομπών, ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται στο πρώτο έγγραφο. Και γι' αυτό θεωρούμε πολύ θετική την πρόταση του εισηγητή. Ως προς το άρθρο 15, κατανοούμε ότι θα πρέπει να οριστούν σαφή κριτήρια για τις εξαιρέσεις, αλλά τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να χάσουμε αυτό το πλαίσιο ευελιξίας που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη και τα περιβαλλοντικά της, ε, με βάση την εντοπιότητα. Άρα στο άρθρο 15 θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή την ευελιξία και ορισμένα επιμέρου σημεία θα μας απασχολήσουν μέσα στις τροπολογίες. Έχει σημασία η συμμετοχή του κοινού στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά έχουμε αρκετές επιφυλάξεις σε σχέση με τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Δεν θα πρέπει να ισχύσει κατά κανόνα να ισχύσει το άρθρο 290, δηλαδή οι πράξεις κατεξουσιοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρώστη δεν είναι εδώ, οπότε ερχόμαστε στον επόμενο μιλητή, πάλι για δύο λεπτά, ο Καρλ Χάις Φλόρενς καταρχήν. Ευχαριστώ. Όταν κοιτούμε το έγγραφο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και βλέπουμε τι έκανε το Συμβούλιο, συγχύζομαι και άκουσα με μεγάλη προσοχή σήμερα όσα ελέγχθησαν και ενευριάζω όλο και περισσότερο έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι όπως και στο Τρίπελ ε, επί χρόνια ζητούσε 10 ε, ε, ε, χιλιόγραμμα από τη μια μεριά και 1,5 από την άλλη. Και τα ίδια κάνει και εδώ. Αν λοιπόν δεν μπορεί να συμμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό εξηγεί γιατί έκανε μία τόσο αντιευρωπαϊκή πρόταση τώρα, διότι η βιομηχανία ζει στη μεγαλύτερη εσωτερική αγορά της Ευρώπης και κατά την πώληση αυτών των προϊόντων όλοι κερδίζουν αλλά υπάρχει και ένα περιβάλλον το οποίο καλύπτει όλους και δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτό μόνο οι ψηλά ιστάμενοι αλλά όλοι και γι' αυτό θα παρακαλούσα να μεταφερθεί αυτό το σχόλιο στον Επίτροπο διότι θα ήθελα να αποσυρθεί αυτή η έκθεση να προταθεί κάτι πραγματικά ευρωπαϊκό διότι έχουμε πολλούς κανόνες με τεράστιες διαφορές. Αυτά δεν μπορεί λοιπόν ε, να ε, παρουσιαστούν σε εθνικό επίπεδο που θα μας ρωτούν σε ποιο επίπεδο συζητάμε, πού ζούμε. Ε, όχι για το Rotary Club ε, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει το έγγραφο αυτό κατά τα άλλα θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε υπό τις συνθήκες αυτές ε, είχα πει ότι θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών και το κάνω τώρα γιατί πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. ο Γέρος Φούσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χέλμουτ Κράμερ για την εξαιρετική έκθεσή του και θα ήθελα να μου επιτρέψει να του πω ότι ζω 30 χρόνια σε μία πόλη όπου μεγάλωσαν και τα παιδιά μου και αυτό, αυτή η πόλη ανήκει σε ε, μία ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γύρω από την πόλη ε, υπάρχουν τέσσερις μεγάλες εγκαταστάσεις ε, καύσεως και ε, γι' αυτό υπάρχει ρήπανση εδώ και 20 χρόνια και συμφωνώ μαζί του ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο καθαρό περιβάλλον. Καταφέραμε όμως να περιμένουμε περιορίσουμε κατά 90% το διοξίδιο του θείου. Παρόλα αυτά όμως δεν έχουμε εξαλείψει όλους τους ρηπαντές. Έχουμε ε, μεν δυνατότητες αλλά στην Τσεχία εξαρτώμαστε από τις εγκαταστάσεις καύσεως άνθρακα και πρέπει να αποφασίσουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε εγκαταστάσεις ε, καύσεως αερίου αν θα βασιστούμε στην ε, Ρωσία για πάροχο της ενέργειας αυτής ή αν θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνική ενέργεια με ε, καθαρές εγκαταστάσεις περιβαλλοντολογικά. Αλλά αυτά θέλουν σκέψη. Θα έπρεπε λοιπόν ε, να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε με το κοινό, να συμμετάσχει και ε, ε, το, η κοινωνία στη συζήτηση αυτή, να γνωρίζουμε αν θέλουν καθαρό αέρα ή αν θέλουν ίσως λίγο πιο βρώμικο αέρα, αλλά διατήρηση των ισχυουσών εγκαταστάσεων, διότι εάν ρωτήσουμε τους ανθρώπους θα σας πούν ότι αν τους κοστίσει λιγότερο καλύτερα να προχωρήσουν έτσι. Ε, ξέρω γιατί ήρθατε με εκπροσώπους της περιφέρειάς σας και μας είπαν τις απόψεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όπως ο κύριος ε, Κράμερ, ε, ο κύριος Κράμερ έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση και θα ήθελα να ενισχύσω την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία έκανε ο Κλάρ Χάιντς Φλόρενς γιατί εδώ εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να διατυπώσουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο και να στηριχθούν οι προσπάθειες του Κοινοβουλίου για να υπάρξει μια καθαρή Ευρώπη διότι η συνθήκη ε, σαφώς υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν έχει φιλόδοξους στόχους και ε, προσπαθεί να κάνει ακόμη περισσότερες τρύπες στο ελβετικό τυρί το οποίο μας έχει παρουσιάσει όπου όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν τις εκπομπές και ε, άρα πρέπει να ισχύσουν και συγκρίσιμες προδιαγραφές για όλους τους Ευρωπαίους. Δεν πρέπει δηλαδή από τη μία πλευρά των συνόρων η μένα είναι πιο φιλόδεξη και η, από την άλλη πλευρά των συνόρων η άλλη λιγότερο. Θα έπρεπε λοιπόν να ε, προσπαθήσουμε να διασώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα από την πρώτη ανάγνωση για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική και να υπάρξει μία κοινή άποψη. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένες ορισμένα δεδομένα αλλά στο, το 15-4 πρέπει να είναι πιο σαφώς διευκρινισμένο να ξέρουμε τι εξαιρέσεις θα υπάρξουν στα κράτη-μέλη γιατί δίδονται οι εξαιρέσεις και τι χρονική διάρκεια θα έχουν διότι διαφορετικά δεν θα λύσουμε τα προβλήματά μας δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι θα βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος με μεγαλύτερη αντιγόνωση. Θα πείτε ότι θα είναι σαν να πείτε ότι θα έχετε καλύτερη ψήξη αν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου σας. Ευχαριστώ. Η Κορίν Λεπάζ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή που όρισε σωστά το ζήτημα. Οι μεγάλες εξαιρέσεις ε, οδήγησαν σε μεγάλη απόκληση των κρατών μελών ως προς τις εκπομπές. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά. Ο κύριος Ζίμπερ είπε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να πλαισιώσουμε καλύτερα τις εξαιρέσεις και να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένας ε, ε, ενδιάμεσος τρόπος ελέγχου των εκπομπών. Το IPPS θα πρέπει να το ορίσουμε καλύτερα και να δούμε κατά πόσο το ΙΠΠΣ τηρεί το περιβάλλον, τις προδιαγραφές του, της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης δεν χρειάζονται εξαιρέσεις για τις ε, μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης μέχρι το 2016 δεν προχωρήσαμε με την ε, οδηγία περί εδάφους. Ο κύριος ε, Κράμερ μίλησε για την ενδεχόμενη χρήση των γεών μελλοντικά. Δηλαδή αν έχει βιομηχανική χρήση τίποτα δεν θα γίνει από τον ε, αρχηγό εκμετάλλευσης, επικεφαλής εκμετάλλευσης. Αυτά. Merci beaucoup. Bogoslav Sonic. Ο Bogoslav Σόνικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκουαρντίνη ο οποίος τόνισε ε, ποιο είναι το πλαίσιο της συζητήσεώς μας, δηλαδή η ε, οικονομική κρίση. Δεδομένης λοιπόν αυτής της κατάστασης θα πρέπει να στηρίξουμε ε, το, την άποψη του Συμβουλίου και να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό. Όσον αφορά τα δύο άρθρα, για το 35 θεωρώ ότι ορισμένες αναλύσεις που θέλουν να βελτιώσουν τις εκπομπές ε, μπορεί να οδηγήσει ε, σε, ε, σε υποβάθμιση των εγκαταστάσεων καύσεως και δεν είναι αυτός ο στόχος μας ε, θέλουμε να υπάρξει μία πολιτική ε, ασφαλείας της ενεργείας και ε, θα πρέπει να υπάρξει μία κατάσταση όπου θα υπάρχει η ασφάλεια αυτή και ε, να υπάρξουν εθνικά προγράμματα. Κανείς δεν θέλει να ζει σε ένα δηλητηριασμένο κόσμο, αλλά πρέπει να δώσουμε χρόνο στα κράτη να επιτύχουν τους στόχους τους. Θα ήταν λοιπόν καλή λύση εάν τα κράτη-μέλη μπορούν να επιτύχουν τους οικολογικούς στόχους, όχι μόνο με αυστηρές προδιαγραφές, αλλά και με μεταβατικές περιόδους για να μπορέσουν να καταρτήσουν προγράμματα τα οποία θα χρειαστούν μία ελάχιστη μεταβατική περίοδο η οποία θα ήταν χρήσιμη. Δηλαδή θα πρέπει να διατηρηθούν αυτές οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νεα κρατη κράτη-μέλη έχουν όντως μια ειδική κατάσταση, το βλέπουμε αυτά. Μάλλον τα νέα κράτη-μέλη έχουν ε, μια ειδική κατάσταση και το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ε, υπάρχουν μεταβατικές περιόδοι, οι οποίες πηγαίνουν έρχονται, είναι ένα επιχείρημα το οποίο προτάσσεται επανειλημμένος και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε μέσα στα πλαίσια του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 poprzez e, e, e, Επιχειρήματά μου ε, ήθελα να σχολιάσω ότι δεν πρέπει να αμφισβητηθούν. Πιστεύω ότι χρειάζεται μία μεταβατική φάση κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα επενδύσεων το οποίο θα επιτύχει τους στόχους τους οποίους επιζητούμε. Δεν προσπαθώ εδώ να καλύψω τους λομπίστες. Ευχαριστώ για τη δήλωση ο Κρίς Ντέιβις. Ο εισηγητής ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος. Υπάρχουν ονειροπόλοι. Εγώ προσπάθησα να το κάνω ακόμα πιο ονειροπόλο τον ε, εισηγητή, αλλά δεν τα κατάφερα. Δύο σημεία ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά πόσο τα ε, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ε, οι υδροηλεκτικές θα μπορέσουν να, να δράσουν για πολλά χρόνια με βάση τις μεγάλες εγκαταστάσεις ε, καύσης. Αυτό αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν έχουν γίνει κατάλληλες επενδύσεις για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων. Γι' αυτή λοιπόν ζητάτε εξαιρέση. Θα πρέπει να μειώσουμε το διεξίδιο του άνθρακα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν για περιορισμένο αριθμό ορών παρά να τις αντικαταστήσουμε με μια νέα γενναία ε, καύσης, ορυκτών καυσίμων. Δεν ξέρω ποιο, είναι οι καλύτερες λύση ποια είναι η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι ομάδες τώρα ως προς τις εκπομπές και τις επιδόσεις. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι το καλύτερο μέσο για μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν να ισχύσουν όταν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη αλλά το πρόγραμμα ανταλλαγής εκπομπών όπως έχει αναδιατυπωθεί σε αυτή την νομοθεσία, δεν επιτρέπει όρια στην εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα τη στιγμή που καλύπτεται η νομοθεσία από το σχέδιο ανταλλαγής εκπομπών. Άρα ο καθένας θα πρέπει να ορίσει στρατηγικές που είναι κατάλληλες για τις ανάγκες του. Γι' αυτό θα χρειάζεται μεγαλύτερη διασάφηση και ελπίζω να δεχτείτε αυτή την κίνηση, την κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Χόλγκερ Κράμερ για την καλή προεργασία που έχει κάνει. Προχωράμε τώρα στο δεύτερο γύρο και όπως είπε στην εισαγωγή τα μεγάλα θέματα είναι οι μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεων όπου θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές. Ευχαριστώ όμως διότι σκέφτηκε και τις μικρές βιομηχανίες και εδώ αναφέρομαι ε, στις μικρές εγκαταστάσεις που επίσης ε, προκαλούν εκπομπές και όπου θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την γεωργία, διότι όσον αφορά τα ε, ε, νητρικά άλατα ε, ξέρουμε την οδηγία η οποία καλύπτει τα απόβλητα της γεωργίας και δεν χρειάζεται να επικαλύψεις αλλά δεν χρειάζεται πάλι να ξανακάνουμε νέες υποδιαιρέσεις για τα πουλερικά παραδείγματος χάρη θα πρέπει να είμαστε συνεπείς δεν πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουμε μία γραμμή η οποία θα οδηγήσει σε κάτι ανόητο. Όσον αφορά τις ε, οριακές τιμές ε, στο παράρτημα 5 ξέρω ότι και εδώ σε ορισμένα σημεία υπάρχουν αντιφατικά ε, απαιτήσει, δηλαδή οι τουρμπίνες αερίου θα πρέπει να μπορέσουν να λειτουργήσουν και με υγρά καύσιμα και την περασμένη χρονιά είδαμε το ε, αποκλεισμό για την παροχή αερίου από τη Ρουσία και δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα ίδια. Υπάρχουν όμως ε, οι οριακές ε, τιμές για τα άλλα τα ζώτου και δεν μπορούμε να τις μειώσουμε παρά μόνο αν έχουμε περισσότερους πόρους από αυτούς που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Μήπως λοιπόν για αυτές τις λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές ε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε μήπως ε, παραλογιζόμαστε στο τέλος. Ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Σκυλακάκης. Κατανοώ ότι ήταν πολύ δύσκολο του έργου του εισηγητή και ήταν δύσκολη οι δύσκολες διαπραγματεύσεις κατά την πρώτη ανάγνωση. Υπάρχουν όμως προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εργαστούμε εις βάθος. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό στη χώρα μου. εχουμε ε, τέσσερις πέντε μονάδες ε, λιγνίτη που θα πρέπει να παροπλιστούν μέχρι το 2020. Εάν περάσει αυτό το σχέδιο θα πρέπει να διαθέσουμε 1,5 δις ε, επενδύσεις για αυτές τις μονάδες που θα πρέπει να παροπλιστούν μέχρι το 2020. Αυτό είναι μεγάλη κατασπατάληση χρημάτων, γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μην γίνονται εξαιρέσεις όταν δεν υπάρχει λόγος, αλλά να βρούμε εκεί που υπάρχουν θεμητά προβλήματα. Και αυτό ισχύει και για τα μικρά νησιά που έχουν διαφορετικές ε, ανάγκες ε, ηλεκτροδότησης τη στιγμή που δεν είναι κανένα συνδεδεμένος με το κεντρικό δίκτυο και για την Ελλάδα ισχύει κάτι τέτοιο όπως και φαντάζομαι σε άλλα κράτη-μέλη. Εκτιμώ τις εργασίες που έχουν γίνει αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει η μεταβατική φάση πιο λεπτομεριακά έτσι ώστε να μην έχουμε κατασπατάληση πόρων και επενδύσεων. Michel Rivasi. Nein, dann Ο äh, Πέτερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, διότι εδώ δεν ομιλώ σαν ε, συντονιστής ε, του περιβάλλοντος και βλέπετε ότι δεν υπάρχει συσπηρωμένη θέση στην πολιτική ομάδα του ΕΛΚ, όπως ε, συμβαίνει και σε άλλες πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα όμως να τονίσω ε, ένα θέμα που έθιξε ο κύριος Κράμερ για την ποιότητα του αέρα. Είναι δικαίωμα του κάθε κράτους και αυτό έχει αποφασιστεί και από το Κοινοβούλιο να επιτύχουν ε, στόχους ποιότητος του αέρα. Και όπως είπε η Ελιζαμπέντα Γαντίνη, έχουμε ακόμη δυνατότητες στον τομέα των μεταφορών και εδώ αντιφάσκω με τον κύριο Κράμερ ε, διότι βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξουν μειώσεις διαφόρων αερίων αλλά όχι μόνο δεν θα επιτύχουμε βελτιώσεις αλλά θα κλείνουν οι δρόμοι και θα κλείνουν περιοχές εάν δεν κάνουμε κάτι και για τους μεγάλους υπευθύνους των εκπομπών διότι δεν θέλουμε μόνο οι μικροί να πληρώσουν το λογαριασμό και ε, να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα λέει «Μα τι αποφασίσατε που οδηγήσω να μου κλείνουν τους δρόμους στη χώρα μου». Εάν λοιπόν θέλουμε μία στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το ψήφισμα το οποίο αποδεχθήκαμε την περασμένη εβδομάδα χρειαζόμαστε μία ε, στρατηγική διαρκείας και γι' αυτό συμφωνώ με όλους όσους λέγουν ότι βεβαίως η Ισπανική Προεδρία πρέπει να κινηθεί. Δεν είναι δυνατόν να λέει ότι δεν διαπραγματευόμαστε με το Κοινοβούλιο πραγμάτευση στη δεύτερη ανάγνωση είναι ο συνήθως τρόπος προόδου. Άρα εδώ πρέπει να ανασκουμποθεί η Ισπανική Προεδρία και να ε, μιλήσει μαζί μας. Η κυρία Χάση. Κάτι το πολύ βασικό, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους του ΕΛΚ, που λένε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί λόγω της παρούσας κατάστασης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κατά την τελευταία θητεία διαπραγματευτήκαμε την νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα και οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ είπανε ότι για να έχουμε πιο αυστηρά κριτήρια για την ποιότητα του αέρα χρειαζόμαστε πρωτογενή νομοθεσία για αυτούς που παράγουν εκπομπές. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με τις πηγές και θα ήθελα οι συνάδελφοι οι οποίοι ζήτησαν αυτή την πρωτογενή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα να είναι συνεπείς. Όταν υπάρχει ακριβώς ε, πρωτογενής νομοθεσία όπως ε, υπάρχει με το IPPC. Και σε σχέση με αυτά που είπε ο Chris Davis ε, για τα, κριτήρια εκπομπών, είδα ότι έχετε το ίδιο, την ίδια ενημέρωση από το WWF. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νομοθεσία έτσι ώστε να μην γίνονται επενδύσεις σε τέτοιες παραδοσιακές μονάδες ηλεκτροδότησης. Ευχαριστώ η Άννα Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να τον συγχαρώ για το σχέδιο έκθεση που μας υπέβαλε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε περί τίνος πρόκειται στην αναθεώρηση αυτή. Πρόκειται να έχουμε ενιαία περιβαλλοντολογικά πρότυπα για καλύτερη προσοχή του περιβάλλοντο και δημόσια υγεία, καλύτερου όρου ανταγωνισμού στην Ευρώπη και αυτό όλοι θα πρέπει να επιτευχθούν με την ενδυνάμωση των βελτίστων ε, πρακτικών και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις πηγές ε, των εκπομπών αυτών, από τις μηχανικές δηλαδή, μονάδες. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν το 2009 ε, ξεκίνησε διαδικασία σε παραβάση για εννέα χώρες μέλη σχετικά με την οδηγία αυτή και σύμφωνα με την ε, περιβαλλοντική υπηρεσία της Κοπενχάγης μόνο τρία κράτη εφαρμόζουν την αρχή της βελτίστης δυνατής πρακτικής. Και παρόλο που έχει λήξει η προθεσμία για την ε, μεταφορά της ε, κοινωτικής οδηγίας σε εθνικό δίκαιο, υπάρχουν 1.500 εγκαταστάσεις ακόμα στην Ευρώπη που δεν τηρούν τις εν λόγω προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες προσαρμογής και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα προβλήματα που έχουμε για τις εκπομπές ε, και οι ποσότητες των εκπομπών είναι από το ένα στο χιλιαπλάσιο σε ορισμένες χώρες και γι' αυτό καλείται η χώρα να, η Κομισιόν συγγνώμη, να ξεκινήσει στις πηγές των εκπομπών αυτών και συμφωνώ βέβαια με τις ε, προδιαγραφές που είχε προβλέψει το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση και που τις ξαναεισαγάγει το, ο εισηγητής μια τελευταία πρόταση για την προστασία των υγεών πρόεδρε. Θα πρέπει να δούμε κάποια λύση για να ξαναεπανέρχουν οι υγείες αυτές στην καλή κατάσταση και όχι στην αρχική κατάσταση. Δεν θέλω να υπάρχει επίσης κανένα προηγούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα 16 τελικά δευτερόλεπτα έγιναν 16, ε, άλλα 16, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Σπινότη. Ευχαριστώ. Η ανάγκη να προχωρήσουμε σημαντικά περισσότερο από την πρόταση είναι προφανές. Θα ήθελα ταυτόχρονα να θέσω ένα άλλο θέμα, το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Και ξέρουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και εδώ ένας από τους στόχους είναι η πράσινη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη εσωτερική αγορά και ισοτιμία στους όρους ανταγωνισμού και θα ήταν πολύ καλό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες μας να είναι ανταγωνιστικές. Αν έχουμε πολύ ε, παρεκκλήσεις και πολύ ε, μακρές περιόδους ε, προσαρμογής, θα έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού και αυτό επίσης δεν βοηθάει την βιομηχανία που θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική και να μεταβιβάσει το κόστος ε, τους πολίτες. Εντάξει, να υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις κάποιες ε, ε, παρεκκλήσεις και υπάρχουν και μεταβικές περίοδοι όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, αλλά από την άλλη μεριά αν είμαστε πολύ επικοί σε αυτά τα δύο σημεία θα είμαστε αντιπαραγωγικοί όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανία μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογο των ομιλητών. Η Μαριάννα Βένινγκ τη Εκκλησική Επιτροπή έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Βένινγκ. Ναι. Καλημέρα σας. Καταρχήν, θα ήθελα να συμφωνήσω με εκείνους οι οποίοι ευχαρίστησαν τον ε, κύριο Κράμερ για την εργασία του και εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εκτίση, αυτή, καλή εξέλιξη σε σχέση με αυτό που είχαμε στην πρώτη ανάγνωση σε πολλά σημεία και πιστεύω ότι από ό,τι ακούσαμε από διάφορους βουλευτές εδώ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. όταν έτσι αυθόρμητα θέλετε να έχετε την αντίρρηση Κομισιόν σε αυτές τις ομιλίες, έχω να πω ότι τα τρία σημεία που συμπεριέλαβε ο κύριος Κράμερ θα μπορούσα ίσως σύντομα να αναφέρω. Καταρχήν έχουμε το δίκτυο ασφαλείας. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις από αυτού. Η Κομισιόν είχε πει ότι υπάρχει αυτή η ιδέα ήδη. Έχουμε ήδη τρεις ή τέσσερις οδηγίες ε, όπου περιλαμβάνουν αυτά τα ελάχιστα πρότυπα μεταξύ αυτών και τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και δεν έχουμε καμία επιφύλαξη εάν πραγματικά χρειαστεί να υπάρχουν αυτά τα ελάχιστα πρότυπα μπορούμε από πλευράς Κομισιόν να τα υποβάλουμε. Το ότι δεν αναφέρονται ε, ρητά στην ε, πρόταση ο οφείλεται στο γεγονό ότι η Κομισιόν έτσι γελώς έχει το δικαίωμα των προτάσεων αυτών. Νομίζω ότι αυτά που προτείνει ο κύριο Κράμερ στην εκθεσή του κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση. Για πρώτη φορά απορρίψαμε την γενικευμένη επιβολή σε όλους τους τομείς για διάφορους λόγους, γιατί πραγματικά πνευματολογικά δεν είναι κάτι τέτοιο λογικό. Εάν τώρα όμως εξετάσουμε τις διάφορες προτάσεις, θεωρούμε ότι ίσως έχουμε τη δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης από το θέματος. Όσον αφορά την ευελιξία, άρθρο 15 παραγραφος 4, είναι ένα σημείο στο οποίο ανέφερθηκαν διάφοροι από τους βουλευτές που πήραν το λόγο και θα έλεγα και για λόγους περιβαλλοντολογικούς αλλά και για λόγους αναγνωστικότητας θα πρέπει να προσπαθήσουμε η πόρτα να μείνει πολύ λίγο ανοιχτή. Υπάρχουν καμιά φορά πραγματικά προβλήματα, αλλά θα πρέπει να περιοριστούμε στην εξαίρεση και η εξαίρεση να μην είναι ο κανόνας τελικά. Τώρα, η συζητήση για πώ θα διατυπώσουμε κάτι τέτοιο στο κείμενο ήταν πολύ αναλυτικέ και εντατικέ και στο Συμβούλιο και θα μπορέσουμε νομίζω να συνεχίσουμε να συζητάμε στο θέμα αυτό για να βρούμε μια αποδεκτή συμβεβαστική λύση. Τελευταίο σημείο, το θέμα των μεγάλων εγκαταστάσεων καύση. Γνωρίζετε τη θέση τη Κομισιόν για το θέμα αυτό. Είχαμε πει ότι είναι αυτός ένας από τους τομείς που πάντα ειστερούσε και για τον οποίο τώρα βελτιώσαμε τα ελάχιστα πρότυπα. Θεωρούμε ότι αυτός ο τομέας δεν θα πρέπει να τύχει διαφορετική μεταχείριση από ό,τι οι άλλοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε όρις εξαίρεσης. Από την άλλη μεριά, σε συζήτηση με το Συμβούλιο είδαμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου. Άρα το να επιμείνουμε στις εξαιρέσεις είναι κάτι που θα πρέπει ακόμα να συζητηθεί. Και πιστεύω ότι η θέση του Κοινοβουλίου γενικά πλησιάζει πάρα πολύ την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Αυτά θέλω να είμαι σύντομη στην αντίδρασή μου. Καταρχήν σας λέω ότι πρόκειται για μια καλή βάση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τον ευκταίο συμβιβασμό μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου όταν άκουσα πολλούς να λένε ότι θα πρέπει αυτό να περάσει στη δεύτερη ανάγνωση, μου φαίνεται ότι αυτό είναι σωστή προσέγγιση και η Κομισιόν θα κάνει οπωσδήποτε ό,τι μπορεί και θα είναι στη διάθεσή σας, θα συζητήσει μαζί σας για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Βένι. Ο Χόλγα Κρέμερ, εισηγητή, έχει την τελευταία λέξη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα είμαι κατά τον σύντομο, γιατί χρησιμοποιήσαμε αρκετό χρόνο. Θέλω να αναφερθώ στο μήνυμα της Άζε Βεσλούν ότι δεν είναι καθόλου θετικό σε σημαντικές συζητήσεις να περιορίζουμε το χρόνο τόσο πολύ. Πολλές φορές συζητάμε μη νομοθετικά κείμενα που θα έπρεπε να είναι μάλλον πίσω-πίσω στην ουρά. Λοιπόν, ο περιορισμό του χρόνου αγόρευση για τόσο δύσκολα νομοθετικά θέματα δεν μου φαίνεται ότι είναι σωστά. Δεν μου φαίνεται ότι είναι καλό αυτό. Θα πρέπει να το ξανασκεφτεί το κοινοβούλιο και να το αλλάξει αυτό. Είδατε αγαπητοί συνάδελφοι ότι εγώ προσπάθησα να πετύχω το τετραγωνισμό του κύκλου με τη λήψη υπόψη των διαφορών τροπολογιών. Δηλαδή αφενός στην κοινή θέση ε, μέχρι το να είναι πιο αυστηρή η έκθεσή μου, άκουσα τα πάντα και κάπου βρέθηκα στη μέση εδώ. Θα πρέπει να κινηθούμε ημέν προς τους δε, εάν θέλουμε να έχουμε κάτι στα χέρια μας στο Συμβούλιο, γιατί στη δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να έχουμε μια σταθισμένη ε, πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι εγώ σας χρειάζομαι όλους και, την κυρία, και τον Μάρτιν Καλεχάν, αν είναι δυνατόν. Θα χαρώ πάρα πολύ να, μας να είμαστε όλοι μαζί. Θα ήθελα να πω πολύ σύντομα κάτι σε ορισμένα σημεία στα οποία μου ζητήθηκε η γνώμη. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει η οικονομική κρίση να ζητηθεί σαν ένα μέσο για να μην προχωρήσουμε. Η οικονομική κρίση πλήττει τους πάντες, κατά νέο τρόπο, και εκείνους που έχουν υψηλά πρότυπα στις ε, βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις. Και γι' αυτό δεν δέχομαι αυτό το επιχείρημα. Ότι δηλαδή χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα οδηγούν σε καλύτερη ανταγωνιστικότητα είναι ασφαλμένο. Γι' αυτό σας ευχαριστώ εσείς που το είπατε αυτό. Δεν θα πρέπει δηλαδή να συγκρίνουμε τους δύο στόχους. Απόδοση στον αφορά το του άνθρακα. Αυτό είναι κάτι που το είχαμε ήδη συζητήσει στην πρώτη ανάγνωση και θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της αποτελεσματικότητας του εμπορίου των εκπομπών. Αλλά όχι μέσα στα πλαίσια αυτού εδώ του νομοθετικού σχεδίου. Γιατί αν επιτρέψουμε αυτή τη σύντηση εδώ, θα αποστρέψουμε το ρωσική από αυτό που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή πώς θα μπορούμε καλύτερα να επιβάλλουμε τη χρήση περιβαλλοντολογικών τεχνολογιών. Γιατί σας το λέω ξεκάθαρα ότι αν αυτό το θέμα του εμπορίου των εκπομπών υπάρχει τελικά στο κείμενό μα, θα έχουμε ακόμη πιο μεγάλα προβλήματα με το Συμβούλιο. Και τέλος. Δύο προτάσεις όσον αφορά το θέμα των συμβιβασμών. Η κυρία Γκαρντίνη είπε ότι αφήνω πολλά περιθώρια κρίση στην Κομισιόν με την έκθεσή μου όταν πρόκειται για τον ορισμό των ελαχίστων προτύπων. Ωραία, ας συζητήσουμε την διαδικασία. Ο Μάρτιν Κανέχαν αναφέρθηκε στην συναπόφαση. Αυτή είναι η πρόταση. Δεύτερη πρόταση. Καταλαβαίνω Ο κύριο Σόνι, τον κύριο Βούσκι που δυστυχώ έφυγε ή εγώ δεν τον βλέπω. Καταλαβαίνω. Ο κύριο και εδώ είναι, ναι, αλλά ο κύριο Ζούσκι δεν είναι εδώ. Τα ίδια επιχειρήματα ακούστηκαν όμω. Καταλαβαίνω, λέω, ότι τα κράτη-μέλη χρειάζονται εθνικά προγράμματα. Εγώ θα μπορούσα να φανταστώ τα προγράμματα αυτά με τροποποιημένη μορφή να τα εντάξουμε στο τέλος στην θέση του Κοινοβουλίου. Αλλά συμφωνήστε μαζί μας για να προχωρήσουμε όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα. Και μια τελευταία τελευταία πρόταση. Η βούληση των κρατών μελών, Καλ Χάιντς Φλόρεντς, δεν φαίνεται να είναι τεράστιο να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα να προστατεύσω λιγάκι και την Κομισιόν, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι παρά τόσο καλή όσο τις επιτρέπουν να είναι τα κράτη-μέλη. Εμείς το κοινοβούλιο, προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την έλλειψη βούληση των κρατών μελών με μια ισχυρή βούληση και θα πρέπει εμείς με τη δεύτερη ανάγνωση να αντιτάξουμε κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να περάσουμε στις διαπραγματεύσεις και με το Συμβούλιο και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα για τη δεύτερη ανάγνωση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Βένιγκ είπε ξεκάθαρα ότι το τροποποιημένο σχέδιο ελεγχής των προτύπων δεν το απορρίπτει πια πλήρως. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας και θα ήθελα να μπορέσουμε στους επόμενους μήνες να εργαστούμε επικοδομητικά για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Πρώτα, σε ευχαριστώ, Χαλκα Κράμερ. Ναι, βρισκόμαστε στη δεύτερη ανάγνωση. Υπάρχουν κάποιες προθεσμίες. Έχουμε το πολύ τέσσερις μήνες ως Κοινοβούλιο μετά την πρόθεση του σκηνιστή του Συμβουλίου. Αυτό έγινε το Μάρτι, την τελευταία σύνοδο. Οι προθεσμίες που θα ακούσετε απορρέουν από αυτά. Η υποβολή τροπολογιών 23 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία 27-28 Μαρτίου στην Επιτροπή μας και μετά τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Είναι στενέ οι προθεσμίε και θα πρέπει λοιπόν να υποβληθούν οι τροπολογίε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημέρα τη διάταξη. Τα πρότυπα επιδόσεων που χωρίζουν από τι εκπομπέ των νέων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Ο εισηγητή μα είναι ο Μάρτιν Κάλαναν. Ευχαριστώ. Περιμένω ένα λεπτό μέχρι ότου επικρατήσει ε, ησυχία ναι, ας περιμένουμε λίγο. The other interest groups have left the room or decide to be silent. Ας περιμένουμε μέχρι να αποχωρήσουν όσοι είναι να αποχωρήσουν ή αν αποφασίσουν να σιωπήσουν, να σιωπήσουν. Okay, I think we continue and those who want to leave the room, please do it silent, then we Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, ας ακούσουμε τον εισηγητή μας, ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Okay, um, CO2 emissions from... Οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα από τα νέα ελαφρά οχήματα. Όσοι ήσασταν ε, στην τελευταία ε, σύνοδο, όπως, ε, όπου μιλήσαμε για, την, ε, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στα ελαφρά οχήματα, θα θεωρήσουν ότι όλα έχουν ήδη υποθεί. Γιατί τα στοιχεία αυτά υπάρχουν και στην πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση ορίζει 157 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα για τα νέα ελαφρά οχήματα που αποτελούν το 10% της αγοράς των μεταφορών. 157 γραμμάρια είναι η πρόταση της Επιτροπής μέχρι το 2014 με ένα phasing in από το 2014 στο 2016. Επίσης προτείνεται προτείνονται και 135 γραμμάρια μέχρι το 2020, μακρόπνος στόχος. Θα θυμόσαστε ότι είχαμε ένα μακροχρόνιο στόχο και σε εκείνη την νομοθεσία. Είναι μια πρόταση που υποστηρίζω. Θα πρέπει να δώσουμε στους κατασκευαστές ε, περισσότερο χρόνο για να ξέρουν ποια όρια απαιτούνται, ποια τεχνολογία θα πρέπει να εισαχθεί και πού πρέπει να βρίσκονται το 2020 ως προς το επίπεδο των, του ορίου. Τα 135 γραμμάρια είναι κάτι το πολύ φιλόδοξο και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή πώς αιτιολογεί αυτό τον αριθμό. Δεν υπάρχουν ε, λεπτομέρειες στη μελέτη αντικτύπου. Φαίνεται ότι λαμβάνουμε υπόψη αυτή την ποσοστή αναλογία και στα μικρά φορτηγά, γιατί η αγορά είναι διαφορετική ως προς τα μικρά φορτηγά. Και η πλειοψηφία της αγοράς κινείται με δίζελ σε σχέση με το πετρέλαιο. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να μας διασαφηνίσει από πού προήλθε αυτός ο στόχος. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν προϋπήρχε ως προς την ε, αρχική διατύπωση είναι τα, η κατακαιρματισμένη αγορά των ελαφρών ε, οχημάτων γιατί πολλοί πολλούν μόνο το σασί και τον κινητήρα. Και υπάρχουν πολλές ε, μήμοι ε, οι οποίες βάζουν άλλα εξαρτήματα σε βαν, σε ψυκτικά οχήματα, σε νοσοκομιακά και ούτω καθεξής. Οι εκπομπές από αυτά τα τελικά οχήματα θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτή την ομοθεσία και δεν έχει νόημα οι ΜΜΕ να είναι υπεύθυνε για αυτές τις εκπομπές. Νομίζω ότι οι αρχικοί κατασκευαστές θα πρέπει να είναι υπόλογοι, αλλά δεν ξέρουμε πώς ε, θα κατανεμηθούν οι ευθύνες. Υπάρχει μια πρόταση στο έγγραφο, η οποία δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. Η Κομισιόν θα πρέπει να μας δώσει ένα νέο non-paper επί του εγγράφου και περισσότερες πληροφορίες ήδη από τώρα. Επίσης υπάρχει μία εξαίρεση για τους μικρούς κατασκευαστές που θα πρέπει να υποστηρίξουμε και να πούμε ότι δεν εξαιρούμε αυτούς τους κατασκευαστές από τις διατάξεις. Απλώς, επειδή έχουν ένα ειδικό output, δεν πρέπει να εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο. Εν πάση περιπτώσει, η πρόταση είναι φιλόδοξη ως προς τα super credits και τις ε, οικολογικές ε, καινοτομίες. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους ε, κατασκευαστές για καινοτομία, για καινοτομίες. Ένα άλλο σημείο που εφήγει είναι να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει ομαδοποίηση του κανονισμού ελαφρών οχημάτων και μικρών φορτηγών ως προς τα επιτρεπόμενα γραμμάρια. Μπορεί να γίνει μια τέτοια ομαδοποίηση, διότι πολλά εμπορικά οχήματα βασίζονται σε ένα γενικότερο αρχικό σχέδιο, άρα μιλάμε για κοινή τεχνολογία. Ως προς το θέμα των κυρώσεων, οι κυρώσεις είναι πολύ μεγάλες για μη συμμόρφωση και άρα οι κατασκευαστές πρέπει να συμμορφωθούν. Θα πρέπει να δούμε όμως το, τις συνολικές γιατί είναι πολύ αυστηρές. Έτσι έχει πρόταση πρόεδρε. Ήρθα σε επαφή με τους άλλους κοιόδης αναμένω τη συνεργασία μας και ελπίζω να φτάσουμε σε μια φιλόδοξη πρόταση και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των άλλων μελών της Επιτροπής σε αυτό το νομοθετικό σχέδιο. Ευχαριστώ κύριε Καλάνα. Ποιος θα ήθελε το λόγο για να κλείσω τον κατάλογο των μελών. Παρακαλώ. Τέσσερα λεπτά για τους ομιλητές και δύο λεπτά για τους υπόλοιπους. Η Άνια Βάσκεβερ είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ για την ε, πολύ καλή παρουσίαση του εισηγητή. Τον ευχαριστώ για τη συνεργασία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια καλή πρόταση. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ε, μια προσπάθεια μειώσεως των εκπομπών και στον τομέα αυτό, δηλαδή των επαγγελματικών οχημάτων κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόκειται για τις ε, συγκοινωνίες, για τις μεταφορές ε, ε, και ήδη έχει προβλεφθεί ότι 15% των εκπομπών οφείλεται εις ε, τα μικρά οχήματα και νομίζω ότι τουλάχιστον καταρχήν είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσο αναφορά τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος ε, έχουμε καταφέρει να τις μειώσουμε κατά 29% μάλλον ο στόχος μας είναι να τις μειώσουμε κατά 29% και ελπίζουμε ότι θα περάσουμε να τον υλοποιήσουμε. Θα πρέπει σε αυτό το τομέα να ασχοληθούμε τώρα με τα επαγγελματικά οχήματα, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Να έχουμε οριακές τιμές οι οποίες να είναι εφαρμόσιμες και να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Γι' αυτό και πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε μία ρύθμιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ε, συνθήκες πλαίσιο διότι ε, αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο κέντρο της πόλεως και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οικονομική κρίση στην οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη ως εκ τούτου δεν πρέπει να ε, δημιουργήσουμε συνθήκες με τις ε, επιταγές μας οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια σημαντική αύξηση των ε, τιμών. Ε, διότι δεν θα επιτύχουμε τον στόχο που επιζητούμε και γι' αυτό ε, εάν κοιτάξουμε και τους αριθμούς ε, όσον αφορά τις εκπομπές των επαγγελματικών οχημάτων έχουν μειωθεί κατά 24% το 2009 και πρέπει να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές αλλά θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για οικολογική καινοτομία και εδώ πάει προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόταση αυτή αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περαιτέρω διότι όπως ελέγχθη υπάρχουν πολλά κοινά σημεία με ε, τα ε, ιδιωτικά αυτοκίνητα και εάν δούμε τι ε, μέτρα είχαμε λάβει τότε πρέπει να δούμε τι μπορεί να εφαρμοστεί για να μεταφερθεί και στα μικρά επαγγελματικά οχήματα και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδείγματο χάρη στο super credits έχει μεταφέρει τις διατάξεις χωρίς να τη στήξει καθόλου, πράγμα το οποίο δεν ισχύει και όσον αφορά τις κυρώσεις δεν έχουν μεταφερθεί ως είχαν, αλλά στα ε, ελαφρά ε, ε, ε, στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το, η υπέρβαση κοστίζει 20 ευρώ ενώ στα ιδιωτικά αυτοκίνητα 95. Πρέπει να συγκρίνουμε συγκρίσιμα πράγματα και ως εκ τούτου η ε, κατανάλωση είναι με ένα ουσιαστικό επιχείρημα και πρέπει να ληφθεί υπόψη και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Ξέρω ότι ο χώρος μου είναι περιορισμένος και θα απαντήσω μόνο σε δύο-τρία σημεία. Δηλαδή νομίζω ότι στις οικολογικές καινοτομίες πρέπει να έχουμε εφικτούς στόχους και όταν κοιτάμε τα, τον τομέα των ιδιωτικών αυτοκινήτων θα πρέπει να σκεφτούμε να δημιουργήσουμε ένα μεταβατικό καθεστώς για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Ο Ματίας ε, ε, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ορισμένα σημεία να ήταν πιο φιλόδοξη, διότι στην έκθεση Σακώνη είδαμε η οποία τώρα έχει αποφασιστεί ότι η βιομηχανία αντέδρασε αμέσως. Έχουμε τα πρώτα μοντέλα ήδη στην αγορά και υπήρξε μία πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βελτίωσε την ε, ε, οδηγία αυτή. Θα ήθελα και στην έκθεση αυτή να είμαστε πιο φιλόδοξοι και θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, διατυπώσει βελτιωτικές να ε, ε, βελτιώσει τις προτάσεις της διότι είναι δυνατόν εάν μειώσει κανείς την ε, ταχύτητα να βελτιώσει τον κινητήρα να μειωθεί η ταχύτητα με την οποία εγχύεται το καύσιμο και άρα να μειωθούν και οι εκπομπές. Άρα θα ήθελα να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η ε, αυτή η πρότασή μου. Βλέπω ότι ο προηγούμενος επίτροπος, ο κύριος Δήμας, δεν είχε υιοθετήσει τις προτάσεις που είχαμε διατυπώσει. Υπάρχει τώρα μία πρωτοβουλία. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόταση, ενώ ορισμένοι την απέφχονται. Αλλά πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε αυτή την οδό θα γίνουμε αναξιόπιστοι. Και αυτό το... Ε, δεν είναι επιθυμητό, γι' αυτό και θα πρέπει αυτή η πρόταση να εφαρμοστεί με φιλόδοξο στόχο διότι ήδη έχουμε ρυθμίσει τον τομέα των ιδιωτικών αυτοκινήτων ο οποίος απεφασίσει στη πρώτη ανάγνωση και άρα ο επόμενος στόχος είναι τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ε, για να μπορέσει κανείς να καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ ε, τους και των ιδιωτικών αυτοκινήτων αυτοκινήτων και ε, ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε στο Κοινοβούλιο. Με ενδιαφέρει πολύ να δούμε ποια θα είναι η επόμενη παρουσίαση. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι διότι με την πίεση υπάρχει καινοτομία και την καινοτομία δεν την βλέπω εδώ στην πρόταση που μας έχει υποβληθεί όσο αναφορά ε, την ε, ε, σκόνη ε, διότι όταν ε, αυξάνεται το βάρος και το φέλιμο βάρος έχει επίσης σημασία θα πρέπει να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αντιμετωπίζει την άνοδο της καμπύλης την οποία είχε διατυπώσει. Νομίζω ότι στο θέμα σακόνη είχαμε μια καλή συμβιβαστική λύση και γι' αυτό την αποδέχομαι ε, όσον αφορά τους στόχους των 175 ε, και 135 γραμμαρίων πιστεύω ότι ο στόχος των 175 γραμμαρίων δεν είναι αρκετά φιλόδοξος διότι ε, υπάρχει ένα face-in το οποίο εφαρμόσαμε και στην έκθεση Σακώνη και θα έπρεπε εδώ το 175 γραμμάρια να αποτελέσει μια οριακή τιμή και στη συνέχεια μπορούμε να προβλέψουμε ότι σε ε, μελλοντικές ε, ε, σκέψεις για το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρουσιαστεί με το πρόσωπο καθαρό, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Τώρα η ο ειδικό μάλλον των εκπομπών, ο Χόλγκερ Κράμερ, είμαι υπεύθυνο των βλαβερών ουσιών στα εργοτάξια, αλλά πιστεύω ότι ο στόχος αυτός είναι αρκετά φιλόδοξος και δεν νομίζω ότι μόνο η ρυθμιστική πίεση δημιουργεί, δημιουργεί την καινοτομία. Η καινοτομία και η βελτίωση μπορεί ε, να δημιουργηθεί και ε, από ανταγωνισμό και γι' αυτό ε, αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία ήδη ελέγχθησαν. Πρέπει να μην ξεχνάμε ο, ποιοι είναι οι λόγοι για την αγορά ενός ελαφρού επαγγελματικού οχήματος ε, που διαφέρει από τους στόχους αγοράς ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου. Δεν ε, ε, είναι ένα, ένας τρόπος προωθήσεως και πιστεύω ότι εδώ η τιμή έχει μεγάλη σημασία και ο, ίσως είναι ο πρώτος λόγος της αγοράς και μετά το θέμα της, ε, της ε, εμφανίσεώς του. Άρα το επίπεδο των εκπομπών είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αγορά. Όσον αφορά την ημερομηνία στόχο δεν πρέπει να, πολύ, να την πολύ συζητήσουμε, να ελπίζουμε απλώς ότι θα εφαρμοστεί και ε, πρέπει να πω ότι το ερώτημα είναι ε, αν το 2010 ο στόχος του 2020 είναι ε, όντως φιλόδοξος, είναι λιγότερο από 10 και μακροπρόθεσμος, διότι εδώ μιλάμε για, για λιγότερο από 10 χρόνια. Πρέπει να μιλήσουμε για μακροπρόθεσμο στόχο. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε πιο ακριβώς. Πρέπει να δούμε πώς θα επιτύχουμε αυτό τον στόχο, διότι αν ε, δεν έχουμε το 2010 οι ηλεκτρικές μεταφορές, μάλλον με συγχωρείτε, το 2020 έκανα λάθος λέει ο μιλητής, ε, το αν δεν έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως το 2020 τότε ενδέχεται αν έχουμε μηχανές εσωτερικής καύσεως να δημιουργήσουμε μία επίπτωση την οποία να απευχόμαστε. Δηλαδή δεν θα μπορούμε πλέον να έχουμε φορτηγά δύο τόνων, θα έχουμε μικρότερα άρα ενός τόνου περισσότερα, θα είναι μικρότερα τα αυτοκίνητα αλλά τα διπλά και αυτό δεν θα οδηγήσει στο στόχο τον οποίο επιζητούμε. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας και να δούμε εάν είμαστε ρεαλιστές επιζητώντας ένα στόχο για το 2020. Ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί είναι σε περίπτωση που δεν ε, σεβόμαστε τις κυρώσεις για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα θα πρέπει να ισχύσουν για τα ελαφρά επαγγελματικά και ε, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη βάση στην οποία βρισκόμαστε αν δεν έχουμε οικοδομήσει το επόμενο σκαλοπάτι. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν υπάρχει επαρκής έλεγχος, δηλαδή εάν πρόκειται για ειδικά αυτοκίνητα, ε, για ε, αυτο, ε, νοσοκομιακά, για αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στην Ήπεθρο, να δούμε τι είναι οι προδιαγραφές οι οποίες χρειάζονται και αν συνάδουν όλα αυτά. Η Σαμπίνε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Οι ε, ε, εκπομπές ε, του Ευρωπαϊκού του ευρωπαϊκού χώρου αυξήθηκαν κατά 36% τα τελευταία χρόνια όπως είπε η κυρία Βάισμπεργκερ ενώ θα μπορούσαν να έχουν μειωθεί κατά 9% τα ε, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ε, ε, έχουν μεγάλη ζήτηση και ε, στο 2007 η κατανάλωση, η εκπομπή του ήταν 2.203 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Γνωρίζουμε ποια είναι η διαδικασία της βελτιώσεως και ξέρουμε πώς μπορούμε να καλύψουμε τα κενά από την οδηγία των ιδιωτικών αυτοκινήτων, άρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και εδώ. Και αν η βιομηχανία λέει ήδη ότι τα μέτρα από την πρόταση είναι πολύ αυστηρά θα έπρεπε να του υπενθυμίσουμε ότι οι τωρινοί στόχοι έχουν αποδυναμωθεί ε, διότι τα 175 ε, γραμμάρια πρέπει από το 2010 να επιτευχθούν το 2016 και οι κατασκευτικές αυτο κινήτων ε, δεν είναι έτοιμοι να μειώσουν τις εκπομπές αν δεν τους δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, ακόμη και αν ε, προσπαθούμε να τους υποχρεώσουμε. Επιπλέον, οι αγοραστές ε, των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων δεν αποφασίζουν τόσο ορθολογιστικά, διότι οικονομικά δεν έχει κανένα νόημα να έχει κανείς πιο ισχυρό κινητήρα αλλά έτσι ε, ε, υπάρχουν οχήματα τα οποία είναι ε, πάρα πολύ ε, γρήγορα και τα φορτηγάκια αυτά συμπεριφέρονται σαν ιδιωτικά αυτοκίνητα, ο οδηγός δεν έχει ειδική άδεια και αυτό μειώνει ακόμη τις δυνατότητες εφαρμογής των βελτιωμένων εκπομπών. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Δεν θα πρέπει ε, μόνο να καθοριστούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, ε, αλλά να προβλέψουμε και έναν βραχυπρόθεσμο στόχο από τον 2012 που να είναι εφικτός. Μπορούν ε, να ισχύσουν να υπάρξουν στην αγορά ε, οχήματα από τη Ρενό και από τη Φόρντο που πλησιάζουν σε εκπομπές των 125 γραμμαρίων το χιλιόμετρο. Δεν νομίζω θα βελτιώσουμε την κατάσταση σε πιο χαμηλά επίπεδα προσπαθούμε ε, να εφαρμόσουμε ε, την οδηγία με στόχο 135 γραμμάρια το 2020 και με μεταβατικές ε, περιόδους εντωμεταξύ. Εδώ οι χώρες δεν συμπεριφέρονται πολύ λογικά και προσπαθούν να σπρώξουν τα πράγματα όσο μπορούν περισσότερο σαν σαν βουλευτήνα της ΓΚΟΕ ε, πιστεύω ότι το 2013 θα πρέπει να ξαναπαρουσιαστεί το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι υπάρχει ο κίνδυνος μια νέα αξιολόγηση θα καθυστερήσει ακόμη την υλοποίηση των στόχων διότι ό,τι αποφασιστεί τώρα δεν πρέπει να αποδυναμωθεί στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για έναν βασικό κανονισμό όταν μιλάμε για το σύνολο του τομέα. Ο εισηγητής είπε ότι είναι 10% του συνολικού τομέα, αλλά θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020 κατά 10% τουλάχιστον και γι' αυτό στις ανταλλαγές αερίων θα πρέπει να κατέλθουμε κατά 15%. Πρόκειται λοιπόν για πολύ ε, σημαντικό στοιχείο. Η αύξηση των πρωτοβουλειών από τον τομέα μεταφορών μας δίνει ένα συν 40% και θα πρέπει να φτάσουμε σε μείον 15% 10% μέχρι το 2002. Ως προς τα μικρά φορτηγά είναι το 12% του στόλου αυτοκινήτων, αλλά έχουμε αύξηση 50% τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μεγάλη αύξηση. Και επίσης η Επιτροπή όταν μιλήσαμε για την ε, νομοθεσία για τα οχήματα μας είπε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αντισταθμίσεις αλλού όπως στα μικρά φορτηγά. Και θα δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές έτσι ώστε να καταχωρούνται τα οχήματα ως μικρά φορτηγά για να έχουν άλλα επίπεδα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δεσμευτικά τα μέτρα όπως ισχύουν για όλα τα οχήματα. Είχαμε μία αύξηση, πρέπει να έχουμε μείωση κατά 40% μέχρι το 2020 γιατί διαφορετικά θα έχουμε 125 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο μέχρι το 2020 δεν είναι πολύ αυστηρός ο στόχος. Όχι, γιατί αν δείτε τα οχήματα της Mercedes-Benz ή της Volkswagen βλέπετε ότι υπάρχει ήδη απόδοση της τάξης 10 ε, με 15%. Γι' αυτό νομίζω τα 125 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο μέχρι το 2020 είναι ένας ε, ευκταίος στόχος. Ευχαριστώ, Ιούντιτ Νέκης. Θα ήθελα να υποστηρίξω τους φιλόδοξους συναδέλφους. Θα πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι και να μην μας πτωίσει η μεγάλη χρηματοοικονομική ε, κρίση σαν δικαιολογία για να μειώσουμε τους στόχους ή να μεταθέσουμε την ημερομηνία θέση σε ισχύ. υποστηριζει τον κύριο Κράμερο όταν είπε ότι το 2020 δεν είναι και τόσο μακρινό και χρειάζεται και μεγαλύτερη προθεσμία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε όλους τους φιλόδοξους στόχους. Επίσης υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι διότι δίνει ένα σχετικό πλεονέκτημα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μιλάμε για περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές μπορούν να εξάγουν οχήματα χαμηλών εκπομπών σε άλλες αγορές, θα μπορούσαμε με αυτή την ευκαιρία να έχουμε πλεονεκτήματα, διότι οι πωλήσει θα διπλασιαστούν ή θα τριπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια. Διαφορετικά άλλοι τομείς θα καταβάλουν το τίμημα. Μιλάμε για μείωση κατά 20-30% και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές σε τομείς που δεν υπάρχουν στο ETS, άρα ο τομέας μεταφορών είναι πολύ σημαντικός. Άρα αν οι μεταφορές ε, δεν τα καταφέρουν, άλλοι πιο αποδοτικοί τομείς θα πρέπει να καταβάλουν το τίμημα, κάτι το οποίο δεν επιτρέπουμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματική και θα ήθελα να φαίνεται από την οδηγία, την εμβέλεια και την προθεσμία ως προς ε, και τα οχήματα και αυτό μέχρι το 2015. Chris Davis. Ο στόχος των ε, μικρών φορτηγών είναι να βοηθήσουν το εμπόριο. Δεν είναι ήδη πολυτελείας. Πρέπει να δούμε πώς θα τους βοηθήσουμε. Το πιο χρήσιμο είναι να λάβουμε μέτρα που θα μειώσουν το κόστος οδήγησης αυτών των μικρών φορτηγών με χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε πολλά λόμπι των αυτοκινητοβιομηχανιών και δεν ακούμε τίποτα από τους χρήστες. Θα πρέπει να αυξήσουμε τους στόχους και να μην παίζουμε με ημερομηνίε και τα σύναφη. Τα 175 γραμμάρια είναι ένας εύκολος στόχος και αυτοί που φτιάχνουν εξαρτήματα μας λένε ότι υπάρχουν ε, τα εξαρτήματα αυτά διαθέσιμα για να έχουμε μειώσεις. Και πολλοί κατασκευαστές έχουν υπερβεί και αυτή τη μείωση ας ορίσουμε 160 γραμμάρια μέχρι το 2016, να μην μιλάμε για 175. Αυτοί που κατασκευάζουν εξαρτήματα λένε ότι μπορεί να γίνει. Ας ξέρουμε από πού προέρχονται τα λόμπι. Όταν είχαμε μια εθελούσια συμφωνία για μείωση εκπομπών, ήταν πολύ λίγα. Το 2005, 2006 και 2007 δεν έγινε τίποτα με τη μειωσή εκπομπών. Στο τέλος η Επιτροπή εισήγαγε νομοθεσία και είχαμε θεαματική διαφορά, διότι άρχισε η αυτοκινητοβιομηχανία να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή ρυθμίσεις, σοβαρές ρυθμίσεις και άρα θα επεργετηθεί ο καταναλωτής λεπτά. Ακριβώς τα δύο λεπτά τηλεόραση. Ο Ρίχαρτ έχει τώρα. Η Κομισιόν με την πρόταση αυτή ακολούθησε την ίδια πρόταση όπως για τα πρότυπα εκπομπών για τα ιδιωτικά οχήματα, παρόλο που υπάρχουν τεράστιες διαφορές καταρχήν όσον αφορά τη χρήση που χρησιμοποιούνται περισσότερο και πιο συχνά από ότι το συνήθες ε, γεωταχή που συνήθως είναι στον καράς και δεν βγαίνει. Επίσης η κατασκευή είναι διαφορετική. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές και εκεί. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες δυνατότητες να δοκιμάσουν κάτι το καινούριο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχάνει το υψηλότερο βάρος. Εκτός αυτού τα επιχειρήματα για την αγορά και χρήση είναι διαφορετικά εδώ από ότι για τα ΙΟΤΑΧΗ. Τέταρτον, δυστυχώς πολλά από αυτά τα οχήματα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ε, ε, εμπλέκονται σε δυστυχήματα. Και αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό πιστεύω ότι η προσέγγιση δεν είναι σωστή να συζητάμε δηλαδή μόνο για τους στόχους ε, του εξωτερικού του άνθρακα. Θα ήταν καλύτερα να υπήρχε μια καινοτομική πρόταση κομισιών. Ε, ώστε η παραγωγή στον τομέα αυτό να μπορούν έτσι να έχουν κάποια κίνητρα για να δοκιμάσουν καινούρια πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι αυτοί έχουν οχήματα τα οποία ε, ε, ε, επειδή χρησιμοποιούνται πολύ είναι πάρα πολύ καλά για τέτοιου είδους δοκιμές. Δεν μπορούμε λοιπόν να συζητάμε για ε, μπαταρίες των 200 κιλών. Νομίζω δηλαδή η προσέγγιση αυτή καθεαυτή είναι υπεραπλουστευμένη και γι' αυτό έχει καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σαν το χάσει. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, the same structures, same arguments. Έχω ε, την αίσθηση του déjà vu. Τα ξαναείδαμε αυτά και λυπούμε που έχουμε τόσες πολλές ε, αποτυχίες στη συμφωνία στο δικτύο του άνθρακα και τόσα πολλά παραθυράκια. Έχουμε ε, ένα facing του 70%, 80%, μετά 100% ελάχιστες κυρώσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα πραγματικό κίνητρο για να βελτιωθεί η τεχνολογία. Και έχουμε και αποκλείσει για μικρούς παραγωγούς. Το πραγματικό θέμα είναι να έχουμε μια πραγματική κατευθυντήρια γραμμή χρονική και όρια δεσμευτικά. Δεν πρέπει να έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά διεθνή ηγεσία. Και αυστηρή στόχη έχουμε ήδη δει ότι είναι η καλύτερη μέθοδος για να ενθαρρύνουμε τεχνολογικές εξελίξεις και να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηγετική στον τομέα της τεχνολογίας. ίσως ε, η λόμπι από την αυτοκυβιομηχανία είναι, εδώ είναι διαφορετική, αλλά όλοι ακούσαμε από την αυτομηχανία ότι τα όρια του διοξιδίου του άνθρακα ήταν πολύ καλά για να προωθήσουν την ε, βιομηχανία να κάνει κάτι. Και τελευταίο σημείο όταν συζητάμε τους μακροπρόθεσμους στόχους. Καλό είναι να έχουμε κάποια προοπτική μακροπρόθεσμη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να έχουμε κάποιους μακροπρόθεσμους στόχους που δεν μπορούν να επιβληθούν, αλλά ε, είναι καλοί όσον αφορά την ιδέα τους πιο σημαντικό είναι ο στόχος του 2020. Ευχαριστώ ο Καλ Χάιντ Φλόρντ, τελευταίο ομιλητή. Αντιθέτως με την IPPC, εδώ ε, το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολούθησε την ίδια οδό και θα ήθελα να τη στηρίξω. Διότι πολλοί λέγουν ότι όλα αυτά τα έχουμε ακούσει ήδη για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα κατά βάση. Δεν έχουν άδικο, αλλά θα ήθελα να τους υπενθυμίσω ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα υπήρχε μία κατάσταση στη Γερμανία ενώ αυτή τη στιγμή ε, έχετε, ε, ε, έχετε μεγάλες βελτιώσεις, δηλαδή ένας κινητήρας 4 ε, λίτρων έχει κατανάλωση 6 λίτρων, οπότε το ότι δεν θα υπάρξει καινοτομία δεν ισχύει στην πρακτική, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να εξηγήσουμε όλα τα προγράμματα για μειώση του διοξιδίου του άνθρακος κατά τους τελευταίους δέκα μήνες. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να εκνευριζόμαστε, διότι όλα αυτά είναι παρελθόν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και στους νεοφερμένους ότι είχαμε τελειώσει το, την συμφωνία το 2007, η οποία εκ των υστέρων κατέρευσε. Ε, ε, ε, πρόκειτο για μια οικειροθελή συμφωνία η οποία μετά κατέρευσε. Άρα πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει δίκιο και η βιομηχανία έχει δίκιο ότι απέτυχε ή στην οδηγία των ιδιωτικών αυτοκινήτων πρέπει να βελτιωθεί εδώ αλλά υπάρχει έχει μία διαφορά με τα φορτηγά και όλα αυτά θα δεν θέλω τώρα να καταναλώνω τον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Από τα λάθη του κανείς μαθαίνει και ε, μπορεί να καταλήξει και σε συμπεράσματα όσον αφορά το μέλλον. Από την Επιτροπή ο Φίλιπ Πόλ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κάλαχαν ε, και τους ομιλητές για τόσες ερωτήσεις. Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και θα προσπαθήσω να απαντήσω τα περισσότερα. Όταν θα έχω δυσκολίες ε, θα δώσω το λόγο ή σε τη συνάδελφό μου. Όπως ξέρετε όλοι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 διατύπωσε μία στρατηγική για να μειώσει τις εκπομπές των μικρών φορτηγών και ε, υπήρξε ε, μία, ε, μία πρώτη συμφωνία τον Απρίλιο πέρυσι και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Εδώ αναφερόμαστε στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα για να καλύψουμε το κενό το οποίο υπήρχε σε αυτή τη στρατηγική. Υπάρχει λοιπόν μία λογική την οποία να ακολουθούμε και, θα το, και το κατάλαβαν και ορισμένοι από τους προλαλήσαντες. Δηλαδή ε, ορισμένα συμπεφωνημένα για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τον σχετικό κανονισμό αντικατοπτρίζονται και εδώ. Ε, ε, βεβαίως υπάρχουν και διαφορές αλλά δεν πρέπει να εκπλησόμαστε. Πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα. Όσον αφορά τους στόχους και την επίτευξη των 135 γραμμαρίων το 2020 περιλαμβάνεται η εξήγηση ή στις, στη μελέτη των επιπτώσεων αλλά ευχαρίστως να το σχολιάσω. Πρόκειται για πολυμορφικά ε, οχήματα όπως παραδείγματο χάρη τα νοσοκομιακά τα οποία όμως δεν καλύπτονται από αυτή, τη ρύθμιση άρα μην φοβάστε το ίδιο δε ισχύει και για τα φορτηγά ψυγεία προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις ε, ειδικές συνθήκες συνθήκες και ε, θα διασφαλίσω ότι η Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα στείλει στην ε, Γραμματεία του Κοινοβουλίου το έγγραφο με τις εξηγήσεις για να μπορέσει να διανεμηθεί. Καθότου είναι ένα στιγμίο που έχει συζητηθεί με τα κράτη-μέλη και μπορούμε ε, να θεωρήσουμε ότι προτείνουμε μία ικανοποιητική λύση. Όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ ε, των ε, κατασκευαστών αυτοκινήτων και κατασκευαστών ε, μικρών φορτηγών. Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν και φορτηγάκια, οπότε εδώ δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς, αλλά μόνο στις εταιρείες οι οποίες παράγουν μόνο επαγγελματικά φορτηγά οχήματα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 και όσον αφορά τις κυρώσεις. Αν είδατε την ε, μελέτη ε, των επιπτώσεων είμαστε σαφείς ε, διότι πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση και γι' αυτό για τα φορτηγά περιλαμβάνουμε 120 ευρώ αντί για τα 95 που προβλέπαμε για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα είναι διαφορετικά και τα υπόλοιπα στοιχεία. Επίσης, τα φορτηγά είναι επαγγελματικά, τα χρησιμοποιούν επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και άλλες. Γι' αυτό είναι καλό να δει κανεί πού βασίζεται αυτή η πρόταση και ε, πώς αντικατοπτρίζεται στην αξιολόγηση των επιπτώσεων. Οι οικονομίες ε, οι οποίες θα αντισταθμίσουν το αρχικό κόστος των οχημάτων θα οδηγήσουν τελικά ε, σε ε, μία ε, οικονομία 2.000 ευρώ δηλαδή θα υπάρξει μία θα υπάρξει ένα στοιχείο και για τον καταναλωτή και επίσης όσον αφορά τα όρια ταχύτητος θα δείτε ότι στα αιτιολογική έκθεση αναφερόμαστε στα όρια ταχύτητος και στο δυνητικό κόστος ή στην εξοικονόμηση που θα απορρέει από τα όρια ταχύτητος. Υπάρχει μειωμένη κατανάλωση καυσίμων και μειωμένες εκπομπές. Όσον αφορά τα 135 γραμμάρια, και ε, τα ε, θέματα μάζας θα ε, δώσω το λόγο στους συναδέλφους, στη συνάδελφό μου. Γιατί πρότεινα τα 155 γραμμάρια. Υπάρχει μία έκθεση με βάση τη μελέτη αντικτύπου για τους μακροχρόνιους στόχους του 2020 και τα 125 γραμμάρια είναι το μέγιστο δυνατό όρο, όριο που αφορά τα ελαφρά οχήματα. Και βεβαίως μιλάμε για τεχνολογίες υψηλού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες. στα 135 γραμμάρια είναι ένας εφικτός στόχος χωρίς να, να έχουμε υβριδιακό ε, στόλο. Μπορούμε να αλλάξουμε τους κινητήρες και οι κατασκευαστές ασχολούνται με αυτές τις επιλογές και εναλλακτικές ήδη από τώρα το 2013 η Κομισιόν θα δει κατά πόσο επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι και τότε θα προετοιμάσουμε μία μελέτη αντικτύπου με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για αυτή την ανάλυση. Τέλος, τα 35 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο είναι ένας παρόμοιος στόχος με εκείνον που υπάρχει στην ομοθεσία μείωσης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό το στόχο, ο οποίος είναι παρόμοιος με αυτό που αφορά τον στόλο οχημάτων γενικότερα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στα μικρά οχήματα και τα μικρά φόρτηγα. Ως προς την αύξηση της ε, ε, μάζας, δηλαδή την αλλαγή διάρθρωσης στο στόλο μικρών φορτηγών θα αλλάξουμε την διατύπωση του παραρτήματος 1 για να δούμε κατά πόσο αυτό το, αυτή η προδιαγραφή αντικατοπτρίζει τη διάρθρωση της αγοράς. Και τη στιγμή που τα μεγάλα οχήματα γίνουν πιο βαρέα, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις οριακές τιμές έτσι ώστε ο μέσος στόχος των 175 γραμμαρίων να τηρηθεί. Σύμφωνα με την τρέχουσα ανάλυση, φαίνεται ότι η αγορά μικρών φορτηγών θα ακολουθήσει μία άλλη εξέλιξη και επειδή υπάρχει μεγαλύτερος εξορθολογισμός θα δούμε την χρησιμότητα των οχημάτων και δεν θα ασχοληθούμε με πολυτελή οχήματα. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αν έχουν άλλο ε, βάρος τα οχήματα αυτά και κατά πόσο θα αλλάξει η χρήση τους. Δηλαδή η αύξηση της ε, μάζας δεν σημαίνει και αύξηση του στόχου, τουλάχιστον στον τομέα των ε, μικρών ε, οχημάτων. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν Κάλαχαν έχει τώρα τον τελευταίο λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τελευταία σχόλια Συμφωνώ με τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από ό,τι άκουσα από την ε, τελευταία προλαλή είπε ότι η αγορά είναι διαφορετική μεταξύ των ιδιωτικών αυτοκινήτων και των φορτηγών. Οι ε, αγοραστές των φορτηγών είναι πιο ορθολογιστικοί, προσέχουν περισσότερο το κόστος και μακροπρόθεσμα ο στόχος τους ε, θα απορρέει από την ρύθμιση για τα αυτοκίνητα. Όσα για αυτά που είπε η κυρία Βάισμπέργερ, συμφωνώ μαζί της, πρέπει να δούμε εάν μπορεί κανείς ε, να αντέξει αυτά τα αυτοκίνητα, διότι δεν έχει, υπάρχει κανένας λόγος να κρατήσει κανείς το παλιό το αυτοκίνητο, εάν ε, είναι απαγορευτική η, ε, η, η, η από τις εκπομπές ε, όλοι θα βγουν χαμένοι και πρέπει να προσέξουμε πόσο μεγάλες θα είναι οι ε, ευκολίες που θα προσφέρουμε. Ε, βεβαίως μου κάνει εντύπωση ότι οι Γερμανοί μιλούν εδώ για όρια ταχύτητος. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι τα σχόλια αυτά θα πρέπει να παρουσιαστούν στις ε, γερμανικές επόμενες εκλογές. Ε, δεν είπα ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη, εξήγησα όμως για, και ήθελα να ξέρω από πού προέρχονταν οι αριθμοί που αναφέρθηκαν. συζητήθηκε η διαφορά μεταξύ των αυτοκινήτων και της, της αγοράς των αυτοκινήτων των ιδιωτικών και ε, των ε, επαγγελματικών οχημάτων. Η αγορά αυτή είναι διαφορετική. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διείσδυση του ντίζελ και υπάρχουν πολύ περισσότερα φορτηγά. Δεν μπορεί δηλαδή να αφαιρέσει όλο το έξτρα βάρος του, του κλιματισμού και άλλων εγκαταστάσεων. Είναι πιο ορθολογιστική αντιμετώπιση. Ε, όσον αφορά τα σχόλια της κυρίας Χάση, δεν συμφωνώ ότι οι υπερβολικές πιστώσεις, οι καινοτομίες είναι μειονέκτημα του, της ρυθμίσεως. Απλούστατα έτσι θα θεσπιστούν και μέτρα που δεν θα θεσπιζόντουσαν διαφορετικά και υπάρχουν ορισμένες καινοτομίες οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές του του περιβάλλοντος ε, ε, όπως το θέμα του φωτισμού που δεν είχαν ληφθεί υπόψη μέχρι τώρα και θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα εις ε, τον κανονισμό για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Άρα νομίζω ότι πρόκειται απλώς για κίνητρα και καλύτερα είναι να χρυσώνει κανείς το χάπι παρά να τρέχει με τη ράβδο. Ε, και ευχαριστώ με τα σχόλια αυτά του Μάρτα Όλαχαν ε, ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση και θα ε, ξανασυναντηθούμε στις 6 Απριλίου στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ.